την έγκριση της ημερήσιας διάταξης για αυτή την εβδομάδα η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του κανονισμού από την διάσκεψη των Προέδρων και την έχετε λάβει. Για σήμερα δεν έχω κάποιο αίτημα αλλαγή. Παρακαλώ. Ζήτησα να παρέμβω για δύο θέματα. Το πρώτο αφορά το άρθρο 163 του κανονισμού για τις παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού. Υπέβαλα πρόταση για να μιλήσω με θέμα τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, τις αποσημειώσεις συγγενών των θυμάτων εκτελεστέντων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Το αίτημά μου απορρίφθηκε διότι ισχυρίζεται η υπηρεσία ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να αναπτύξω τις απόψεις μου όμως κύριε πρόεδρε βλέπω για πρώτη φορά να μην γίνεται η συζήτηση δευτέρα όποτε πάντοτε έμπαινε η συζήτηση για τις παρεμβάσεις ενός λεπτού και έχει προσδιοριστεί για την πέμπτη όπου την πέμπτη έχουμε μόνο δύο ώρες για το θέμα αυτό και για πολλά άλλα ζητήματα. Εάν όμως κύριε Πρόεδρε, okay, εάν όμως, κύριε Πρόεδρε είχε τεθεί το θέμα σήμερα Δευτέρα που τελειώνουμε στις 7 η ώρα θα μπορούσε να πάμε μέχρι τις 10 και τις 11. Διότι κύριε Πρόεδρε το δικαίωμά μας να μιλήσουμε κάθε φορά δεν μπορεί να εξαρτάται από τον περιορισμό του χρόνου. Και σας ζητώ λοιπόν να προσδιορίσετε το θέμα αυτό για τη Δευτέρα σήμερα, ούτω ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε όλοι οι βουλευτές. Διαφορετικά κύριε Πρόεδρε, παραβιάζεται το δικαίωμά μας. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ήταν σαφές αυτό το οποίο είπατε. Πρώτα απ' όλα ε, αλλαγές ε, τέτοιες αιτήματα για αλλαγές ε, τέτοιας φύσης πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 4 η ώρα. Επειδή είστε νέος βουλευτής σας το λέω αλλά δεκτώ το αίτημά σας. Η αναβολή όμως δεν έγινε για καθαρά τυπικούς λόγους. Έχουμε ακροάσεις απόψε για την στελέχωση δύο θέσεων επιτρόπων. Γι' αυτό το λόγο όλος εξαιρετικός οι ομιλίες του ενός λεπτού μετατέθηκαν σε άλλη μέρα. Γιατί ακριβώς ε, έπρεπε να προβλέψουμε χρόνο και χώρο βεβαίως και παρουσία των βουλευτών για τις ακροάσεις. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι το ουσιαστικό και καθόλου τυπικό. κυρία Φων Στόρχ, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα, τουλάχιστον στη γερμανική μετάφραση. Τετάρτη 12 η ώρα μας λέτε εκλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται προφανώς για λάθος. Δείτε το και στις άλλες γλώσσες, γιατί στο άρθρο 17, παράγραφος 7 της συνθήκης αναφέρεται ρητός πως οι εθνικές κυβερνήσεις επιλέγουν τους εκπροσώπους τους για την Κομισιόν. Και το Κοινοβούλιο μπορεί μόνο να ψηφίσει ενσώματι τους 28. Σας παρακαλώ λοιπόν να διορθώσετε τη λάθος διατύπωση που υπάρχει στην μερίσια διάταξη. Ευχαριστώ. Das ist äh, sicher Μάλιστα ενδιαφέρον και αυτό. Το άρθρο 118 του κανονισμού ε, προβλέπει πως ε, ψηφίζεται από το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, παρότι νέος βουλευτής γνωρίζω ότι το αίτημα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 4 η ώρα. Από τις 11 το πρωί αναζητώ στο τηλέφωνο της υπηρεσίας σας και δεν έχω βρει κανέναν για να θέσω το θέμα αυτό. Είμαι εδώ το δεύτερο λοιπόν θέμα που θέτω κύριε πρόεδρε αφορά στο κατεπήγον. Αυτή τη είχε τεθεί μια πρόταση να συζητηθεί ως κατεπήγον το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό απερίφθη από το Προεδρείο. Όμως σήμερα ήδη τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος έχει εισέλθει στην ΑΟΣ και δημιουργεί προβλήματα. Ζητώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε εδώ στην Ολομέλεια να πάρουμε απόφαση να συζητήσουμε αυτό το κατεπήγον θέμα διότι είναι καθοριστικό για τη διατήρηση της ειρήνης okay, το κατάλαβα αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν έχει ούτε μία σχέση με την ε, ημερήσια διάταξη. Τώρα τι να σας πω, αν δεν τους βρήκατε στο τηλέφωνο υπάρχει υποδομή, μπορείτε να στείλετε ένα email το οποίο θα απαντηθεί αμέσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην Τρίτη. Όχι, ακόμα στη Δευτέρα είμαστε. Δευτέρα, για τη Δευτέρα θέλετε να πείτε κάτι. Για τη σημερινή ημερήσια διάταξη ή για κάποια άλλη μέρα. Τη Δευτέρα είμαστε, αγαπητέ κύριε, στην ημερήσια διάταξη της Δευτέρας. Ζητάτε το λόγο για Δευτέρα ή άλλη μέρα. Την Τρίτη. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στην Τρίτη. Σας παρακαλώ αγαπητέ συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη των Προέδρων προέβλεψε να καλέσει για τη συζήτηση για τα δημοσιονομικά πρώτον το θέμα του προσχεδίου για το 2015 και δεύτερον τον δεύτερο διορθωτικό για το 2014. Συμφωνώντας με το σύνολο των συντονιστών της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα ήθελα να αντιστρέψουμε την σειρά της συζήτησης. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον διορθωτικό του 2014 και στη συνέχεια με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015. Στην πραγματικότητα η συζήτηση θα αφορά τα 300 δις του προγράμματος Juncker, αλλά προς το παρόν το βασικό αντικείμενο της δημοσιονομικής συζήτησης είναι το θέμα των μη καλυμμένων υποχρεώσεων γιατί από το 2010 βλέπουμε ένα ποσό το οποίο δεν καλύπτεται και μεγαλώνει. 5 δις το 10, 11 το 11, 16 δις το 12, 23 το 13 και ίσως το τέλος του 14 να φτάσουμε στα 30 δις. Μιλάμε για ένα χρέος ύπουλο και δεν μπορούμε εμείς να αλλοιώσουμε τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές αγνοώντας τις και αφήνοντας απλήρωτες αυτές τις υποχρεώσεις, ακάλυπτες αυτές τις υποχρεώσεις. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον διορθωτικό του 14 είναι θα έλεγα μια ευκαιρία σταθεροποίησης αυτού του χρέους. Ο τριμερής διάλογος που έγινε την προηγούμενη πέμπτη μας έδωσε τη δυνατότητα να θέσουμε την πρόταση αυτή όλοι οι συντονιστές. Πρώτα ο διορθωτικός του 14 και μετά ο προϋπολογισμός του 2015. Γι' αυτό λοιπόν να μιλήσουμε την Τρίτη και την Τετάρτη με διαφορετική σειρά τα θέματα αυτά. Ξανά τα λέω. Πρώτα ο διορθωτικός του 14 και μετά ο κανονικός του 2015. Σας ευχαριστώ κύριε Τουή. Από αυτό αποφασίστηκε σε συμφωνία με τις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες στην διάσκεψη των πρόεδρων και είπαμε πως ο διορθωτικός προϋπολογισμός 2 του 2014 θα έρθει πιο μπροστά και θα συζητηθεί πριν από τον γενικό προϋπολογισμό του έτους 2015. Οπότε ε, ήδη έχει γίνει αυτό το οποίο ζητάτε. Επίσης, σας ευχαριστώ ε, για το ότι ενημερώνεστε για τα γεγονότα γιατί εμείς ε, δυστυχώς ε, τα προηγούμενα χρόνια με τον προκάτοχό σας ε, φέρναμε πάντα πιο νωρίς τους διορθωτικούς προπολογισμούς. Λοιπόν, για την τρίτη υπάρχει τίποτα, όχι, τετάρτη η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών ζήτησε δήλωση της ε, είπα της εκπροσώπου για την θανατική ποινή για την ε, Άζια Μπίμπη την Τετάρτη ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη χωρίς συζήτηση. Ο κύριος Φαντάλεν έχει το λόγο από αυτού. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν μιλάω μόνο εξ ονόματος της ομάδας μου, αλλά και ως συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας για την ελευθερία της πίστης του Κοινοβουλίου. Ως ομάδα εργασίας, κύριε Πρόεδρε, είμαστε κατά της νομοθεσίας της βλαφημίας του Πακιστάν, με βάση την οποία μπορεί ο κόσμος να καταδικαστεί ε, αν προσβάλλει τον προφήτη με υψηλότερη προβλεπόμενη ποινή την θανατική ποινή όπως ε, όντως καταδικάστηκε η Άζια Μπίμπη σε θάνατο για βλασφημία. Είχε αναφερθεί μάλιστα νομίζω από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ρητός ε, η κυρία αυτή την ε, δε Πέμπτη την οποία μας ε, πέρασε ένα δικαστήριο στην Λαχώρη επιβεβαίωσε την καταδίκη της ε, κυρίας Μπίμπη οπότε τώρα θα πρέπει να προλάβουμε την εκτέλεσή της και να ζητήσουμε να αλλάξει αυτή η νομοθεσία περί βλασιμίας. Αυτό ακριβώς θα θέλαμε να ακούσουμε από την κυρία Ήπατη εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ. Für den Antrag möchte Frau ε, Κυρία Μπιόρκ θέλει να τοποθετηθεί από αυτό. Υπέρ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ΓΚΟΕ ενδιαφερόμαστε πολύ για αυτή την περίπτωση αλλά διαπιστώνουμε επίσης ότι αυξάνονται οι θανατικές οι θανατώσεις. Είναι πολλοί αυτοί που εκτελέστηκαν, που τους επιβλήθηκε η θανατική ποινή και εκτός από αυτή την κυρία και άλλοι πολλοί και ακόμη άλλοι παραμένουν την εκτέλεσή τους πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα ως προς την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και για τη θανατική ποινή θα ήθελε κάποιος να μιλήσει κατά αυτού του αιτήματος κατά όχι, αν είναι κάποιο κατά. Οπότε θα το ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ για να μπει ω τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, διανατάσσεω χειρός. Κατά. αποχέ. Ωραία, εγκρίνεται. Δεν έχω άλλα αιτήματα για την, την Τετάρτη. Για την Πέμπτη. Υπάρχει κάτι. Όχι. Για την πέμπτη. Παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα τι βάλαμε στην ημερήσια διάταξη. Υπήρξε μία πρόταση και μία αντιπρόταση από δύο ομάδες. Έγινε μία ψηφοφορία, δεν κατάλαβα καλά. Τι ακριβώς ψηφίσαμε να μπει στην ημερήσια διάταξη. Το αίτημα του κυρίου Φαντάλεν προέβλεπε η κυρία Άστον στην δήλωσή της να ε, περιληφθεί εδώ πέρα ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένα ε, μία δήλωση για την ε, κυρία Μπίμπη. Η κυρία Μπιόρκ του υποστήριξε και δεν μίλησε κανείς κατά αυτού του αιτήματος. Η κυρία Μπιόρκ μίλησε Μα ρώτησα ποιος υποστηρίζει αυτό το αίτημα και εκεί πέρα ζητήσατε το λόγο. Είπατε πως θέλετε μια ευρύτερη συζήτηση. Μια ευρύτερη συζήτηση από μια δήλωση της υπάτης εκπροσώπου. Από Μα δεν υπάρχει κάτι το ευρύτερο. Παρακαλώ πείτε μας, ναι. Κοιτάξτε, εγώ ζήτησα αντί να μιλήσουμε για μία συγκεκριμένη περίπτωση να μιλήσουμε για το ευρύτερο θέμα της θανατικής ποινής. Να μην περιοριστούμε μόνο σε μία περίπτωση αλλά να εξετάσουμε το σύνολο του φαινομένου των θανατικών καταδικών που αυξάνονται παγκοσμίως. Μάλιστα, τώρα το κατάλαβα κάπως καλύτερα. Είχα καταλάβει πως παρόλα αυτά, γιατί ζητήσατε το λόγο όταν είπα ποιος είναι υπέρ αυτού του αιτήματο. Ε, και πράγματι επί της αρχής δεν στηρίζεται αυτό το αίτημα, είναι μια αναλλακτική πρόταση. Αλλά ε, είχα την εντύπωση, νομίζω από την ψηφοφορία, πως η συντηρητική πλειοψηφία είναι υπέρ του αιτήματο Φαντάλεν. Οπότε πράγματι ε, ακούσαμε αυτό το οποίο είπατε, το οποίο θα ληφθεί υπόψη για μια ευρύτερη συζήτηση για την ε, θανατική ποινή. Αλλά νομίζω πως υπήρξε ευρύτατη πλειοψηφία για το αίτημα του κυρίου Φανταλεκτός. Αν θέλετε να ξαναψηφίσουμε αν επιμένετε για το δικό σας. Αυτό, αυτό είπα. Περιμένετε να ακούσετε ολόκληρη τη μετάφραση και μετά. Οπότε, κυρία Μπιόκ, θέλετε να ψηφίσουμε το έτοιμά σας. Ωραία. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Το ε, εναλλακτικό αίτημα είναι αυτό της κυρίας Μπιόκ. Να μην μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να έχουμε μια γενική συζήτηση για τη θανατική ποινή. Όποιος είναι υπέρ παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στο... Να ξανα... Περνάμε στο αίτημα του κυρίου Φαντάλεν. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Σαφώς η πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για την πέμπτη υπάρχει τίποτα άλλο. Όχι. Περνάμε τώρα στην δήλωση της Κομισιόν καλύτερη πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον λόγο έχει ο κύριος Μπόργο, ο Επίτροπος Μπόργο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της